I think there limits uh, for those who have come in terms of waiting for the others. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκεί, περιμέναμε όσο γινόταν τους άλλους, να ξεκινήσουμε όμως τώρα με το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη που είναι το σχέδιο έκθεσης του κύριου Ανδρέα Κοτσολίνο για την αστική ανάπλαση ως συμβουλή στην οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Κύριε Κοτσολίνο, έχετε το λόγο. Sí. Eh, molto rapidamente. Eh, Πολύ σύντομα. Η ιστορία της Ευρώπης είναι η ιστορία των πόλεων της. Και η πόλη είναι ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σήμερα στις πόλεις ε, ζουν γύρω στα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελούν ε, το, τη σκηνή για το, τις πιο σημαντικές και οξύες οικονομικές και κοινωνικές συγκρούσεις, αλλά επίσης είναι το πεδίο ευκαιριών ε, είναι οι πόλεις οι οποίες ε, διαρκώς αντιμετωπίζουν τις κρίσεις τις κρατικές και η Ευρώπη χρειάζεται να έχει μια αστική πολιτική, μια πολιτική για τις πόλεις τα κέντρα. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Δεν υπάρχει νομική βάση για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα αξιοποίησης και ανάκαμψης των πόλεων στην Ευρώπη. Ούτε έχουμε μια πολιτική για τη χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας ε, με στόχο της πόλης. Οπότε το θέμα που θέτουμε με αυτή την έκθεση είναι ακριβώς το θέμα της συνέχειας και του εντοπισμού μιας νομικής βάσης ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική προς τις ε, πόλεις και τις, ε, τα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που εγώ προτείνω. Να δοθεί συνέχεια στην εργασία μας αυτή, να δώσουμε μέλλον σε αυτή την πολιτική και αν ε, την θεωρούμε όντως ε, καθοριστική σημασία για την Ευρώπη. Έπειτα, μαζί με το θέμα των πόλων υπάρχει και το θέμα της ε, αναβάθμισης των πόλεων πολιτικές διάφορες έχουμε δοκιμάσει σε διάφορες εποχές και σε διάφορες ε, φάσεις. Ωστόσο, φτάσαμε σε ένα σημείο που χρειάζεται πλέον να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Υπάρχει το σημαντικό θέμα της ε, διάχυτης δυσαρέσκειας και έλλειψης ε, ε, καταλημάτων, το θέμα της ανάγκης να υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερα άελα και υλικά αγαθά που θα πρέπει να υπάρχουν στις πόλεις μας. Το θέμα γενικά της αναβάθμισης των αστικών κέντρων, το μέγα θέμα των περιφερειών των μεγάλων ε, πόλεων όπου συχνά η ποιότητα ζωής είναι πολύ χαμηλή και εκεί εστιάζονται και πιο οξύες ε, αντιφάσεις κοινωνικού τύπου στην σημερινή Ευρώπη. Και έτσι το θέμα της ε, αναβάθμισης των αστικών κέντρων θα πρέπει να αποτελέσει ένα, μια από τις βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της Ένωση. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τις υποδομές, ε, τις ε, σιδηροδρομικές, τις οδικές, τις ψηφιακές. Είναι τρομερές αυτές οι υποδομές και θα έπρεπε υπό το φως όλων αυτών των προβληματισμών να έχουμε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης και αναβάθμισης ευρωπαϊκού χαρακτήρα για τις πόλεις. Ακόμα και ο πειραματισμός με, με, διάφορους, με διάφορα δημοσιονομικά μέτρα, όπως ας πούμε τα ομόλογα έργου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις πόλεις, τα αστικά κέντρα. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, έχουμε το θέμα του εντοπισμού μιας νομικής βάσης που θα δώσει προοπτική και συνέχεια στο θέμα των αστικών κέντρων. Έπειτα, ε, θα πρέπει να έχουμε το θέμα της ε, αναβάθμισης των αστικών κέντρων ως ένα βασικό στόχο ανάκαμψης και αναβάθμισης. Επίσης, ως επίκεντρο της πολιτικής ανάπτυξης και σε αντίθεση με την ε, κρίση στην οποία έχουμε βυθιστεί εδώ και κάποια χρόνια. Το θέμα λοιπόν αυτό θέτει ένα, το θέμα της ανάπτυξης το οποίο δεν θα στηρίζεται μόνο σε ε, φούσκες ε, του οικοδομικού τομέα, του κατασκευαστικού τομέα όπως τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα οικονομική και κοινωνική ένα μέγα πλάνο, ένα μέγα σχέδιο για την αναβάθμιση των αστικών κέντρων σημαίνει σωστή απασχόληση σωστή απασχόληση και κυρίως για τους νέους. Σε αυτά βασίζεται λοιπόν η έκθεση. Αυτή είναι η αιτιολόγηση και εύχομαι να μην αποτελέσει απλά ένα φωτεινό ε, παράδειγμα το οποίο μετά θα εξαφανιστεί, να μην είναι ένας διάτοντας αστέρας, αλλά ότι θα δοθεί συνέχεια έτσι ώστε να αναβαθμιστούν όντως τα αστικά κέντρα. Σας ευχαριστώ. Η Μιλία Ματζόνη δεν είναι εδώ, η κυρία Μανέσκου δεν είναι εδώ, η Καρίμα Νταλή, Ντελή είναι εδώ όμως, έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την παρουσίαση. Εδώ είμαι. Είναι θέματα που ξέρουμε θα πάρουν όλο και μεγαλύτερη διάσταση στο μέλλον δεν έχουμε σχέδιο μπροστά μας προς το παρόν για την έκθεση αυτή και είναι δύσκολο να κατάσουμε τροπολογίες. Αλλά να υπενθυμίσω όταν μιλάμε για αυτή τη διάσταση για την, ε, ε, το θέμα μας πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα σχετικά προβλήματα με την περιφέρεια και την Ήπεθρο. Υπάρχει γυτνίαση και εμείς οικοδομούμε ε, την κατάσταση του 21ου αιώνα και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, αποφεύγουμε να κάνουμε μια, ένα ανταγωνισμό ανάμεσα στο αστικό και μη αστικό περιβάλλον. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο εγώ δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα χαρώ να συμβάλλω όσο μπορώ στην εργασία του εισηγητή με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ε, I understand Cornelia... Η Κορνέλια είναι εδώ. Μπλάσακ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν, και εγώ θα ήθελα να πω ότι το θέμα είναι ύψης της σημασίας θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι πόλεις και τα αστικά κέντρα ως μέσα ανάπτυξης και να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσουν οι πόλεις μας. Ως προς τις ε, οικονομίες μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας από τις ε, πόλεις ε, μέσω ε, μεταφορών μέσω θέρμανσης ή ηλεκτρισμού. Θα πρέπει να είναι μέσα φιλικά προς το χρήστη και δεν μπορούμε να εργαστούμε ανεξάρτητα από τους καταναλωτές ή εθνικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τις πόλεις και τις κομοπόλεις και οι λεγόμενες τηλεπόλεις η, τα δημαρχία, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλα αυτά είναι φορείς ε, συνεργασίας. Ως προς το μέλλον, μέσω διαρθρωτικών ταμείων και ταμείου συνοχής, θα ήθελα να πω επ' αυτού ότι οι πόλεις είναι αυτές που ορίζουν τις προτεραιότητες. Thank you very much. Ε, marie Sanchez. marie Sanchez. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, ΣΥΤΗ. Θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι έχουμε να ακούμε με ένα θέμα που αφορά την αναδιαμόρφωση του ε, περιβάλλοντος στην περιφέρεια. Έχει μια οικονομική διάσταση αυτό και εδώ έχουμε να κάνουμε αποφάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν για την οικονομική ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πραγματικά να το έχουμε στο μυαλό μας και προτάσεις και αυτά που ανέφερε ο συνάδελφός μας, εγώ συμφωνώ, διότι ανέφερε για τις δράσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε χώρες που υπάρχουν ήδη, ε, συνεργασίες ανάμεσα σε πόλεις, κοινότητες. Εμείς ίσως να τις ε, θεωρήσουμε σε ευρύτερες, ε, <clears throat> θα λέγαμε, αστικές περιφέρειες. θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη διότι είναι αυτές οι συνεργασίες οι οποίες έχουν γνώση, έχουν εμπειρία και μπορούν να συμβάλλουν. Και να πω και στον εισηγητή διότι ανέφερε κάτι για νομική βάση. Μήπως θα μπορούσε να το διευκρινίσει αυτό, να το κάνει πιο συγκεκριμένο. Τι υπάρχει πίσω από αυτή τη θέληση να εξασφαλίσουμε και μια νομική βάση. Νίκος Κύριος Χρυσόγελος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα η παρέμβαση της πόλης ε, μπορεί να έχει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, σε μια εποχή ιδιαίτερα σαν τη σημερινή που η κρίση είναι πολύ μεγάλη έχουμε τις πόλεις να υποβαθμίζονται σε μερικές περιοχές ενώ σε άλλες περιοχές έχουν δείξει παραδείγματα ανάκαμψης. Και έτσι θα, πρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική ώστε οι πόλεις συνολικά στην Ευρώπη να ανακάμψουν περιβαλλοντικά αλλά και να πετύχουμε στόχους κοινωνικής συνοχής. Η οι επενδύσεις στα θέματα της ε, αναγέννησης των πόλεων μπορούν να προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας αλλά πρέπει να το δούμε και πώς θα μετέχουν με έναν πιο ευέλικτο τρόπο οι τοπικές κοινωνίες σε κάτι τέτοιο. Μπορεί να δημιουργηθούν ε, μορφές οικονομικής δραστηριότητας που είναι πιο βιώσιμες. Έτσι θα πετύχουμε, εάν έχουμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο, και να μειώσουμε τα αέρια ε, που αλλάζουν το κλίμα, την εκπομπή αερίων που αλλάζουν το κλίμα, να πετύχουμε σε θέματα κοινωνικής συνοχής και να πετύχουμε και σε θέματα ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πόλεις είναι σήμερα αυτές που υποφέρουν κατά πολύ από τα θέματα της ανεργίας και της φτώχειας. Ειδικά στον Νότο, στις χώρες που περνάνε σήμερα μια βαθιά κρίση, αυτό είναι πολύ έντονο. Όταν ένας στους δύο νέους είναι σήμερα άνεργοι και όταν τα ποστά ανεργία στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουν ξεπεράσει το 22%, 23%. Έχουμε φαινόμενα πραγματικά κοινωνικής κατάρρευσης στον ιστό των πόλεων. Και βέβαια αυτό οδηγεί και σε αύξηση εγκληματικότητας και της ξενοφοβίας. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι πρέπει να, εκτός από τα γενικά σχέδια που θα έχουν και επιστημονική και τεχνοκρατική διάσταση, πρέπει να δούμε και τα θέματα δημοκρατικού σχεδιασμού. Δηλαδή πρέπει οι πολίτες να έχουν ε, να συμμετάσχουν ενεργά στο να διαμορφώσουν από κοινού με τους τεχνοκράτες, με τους ε, επιστήμονες το πώς θα εξελιχθούν οι πόλεις τους. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στα σχέδια αναβάθμισης των πόλεων, να μην απλώς θέματα real estate και θα πρέπει να βρούμε και ευέλικτα συστήματα χρηματοδότησης γιατί σήμερα ξέρουμε ότι μερικές φορές υπάρχουν χρηματοδοτήσεις κυρίως μέσω συστημάτων με τις τράπεζες αλλά τελικά αυτές δεν αξιοποιούνται έτσι όπως ε, ε, είναι σήμερα οι συνθήκες λόγω κρίσης. Άρα πρέπει να βρούμε σχήματα ευέλικτα για χρηματοδότηση στα οποία να μπορούν να επιφωληθούν και οι πολίτες άμεσα και εύκολα σε μια εποχή που δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα προκαταβολικά και να περιμένουν πολύ καιρό για να πάρουν πίσω οποιασδήποτε επενδύσεις. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα δούμε μέσα σε ένα ενιαίο σχέδιο ε, που αφορά την αναγέννηση και αναβάθμιση των πόλεων με οικολογικά χαρακτηριστικά αλλά και με κοινωνικά χαρακτηριστικά για πετύχουμε αυτό που θέλουμε βέβαια τα θέματα της κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο για το θέμα των αστικών κέντρων. Γιάν, όχι. Ωραία, λοιπόν. Από την Κομισιόν υπάρχουν κάποια σχόλια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Μόνο μερικά σχόλια η Κομισιόν καλωσορίζει αυτή την πρωτοβουλία και συμμερίζεται τις παρατηρήσεις που αναφέρονται εδώ και τονίζει ότι κάποιες από αυτές είναι βασικές και κύριες αρχές ε, επί των οποίων ε, στηρίζεται η στήριξη των πόλων μέσω του ERDF. Είναι το, η βάση για την συμμετοχική προσέγγιση στα διάφορα επίπεδα δηλαδή της διοίκησης και τους πολίτες. Η Κομισιόν έχει μια μακρά παράδοση δραστηριότητας στο πεδίο της ανάπτυξης των αστικών κέντρων και παρότι ότι η αστική πολιτική η ίδια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα τελευταία 20 χρόνια μια κοινή μεθοδολογία αστικής ανάπτυξης έχει εξελιχθεί και επίσης έχουν αναπτυχθεί στρατηγικές για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Έχουμε το πιλωτικό πρόγραμμα Urban το οποίο ακολουθήθηκε από δύο προγράμματα ακόμα αστικών, ε, μάλλον ε, προγραμμάτων κοινοτικών Urban που οδήγησαν σε πολλά προγράμματα ακόμα στην ε, σημερινή προγραμματική περίοδο. Για το μέλλον, ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης Urban είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020. Ε, θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία θεωρείτε σκόπιμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Σαντιάγο. Δεν ξέρω αν η κυρία Ματσόνη θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, γιατί έχουμε ακόμα πέντε λεπτάκια. Eh, ε, μέσα σε ένα λεπτό θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι αυτή η πρόταση ψηφίσματος είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Μιλάμε για διεξοδική απαρίθμηση όλων των μέσων στην πρόταση ψηφίσματος. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία υπόδειξη στον εισηγητή ε, εν είδη τροπολογίας θα εξαρτήθει πώς θα αντιμετωπίσει του σκιώδης. Πρόκειται για μία ανατροπή του τελευταίου τμήματος, διότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε την πράσινη διάσταση και την έννοια της οικοσυμβατότητας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα του συστήματος αποκομιδής της πόλης. Θα ήταν σκόπιμο να προβάλλουμε αυτό το μήνυμα και κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα οι πόλεις να αναφέρονται ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη γενικότερα και την προώθηση δράσεων για την έξοδο από την κρίση, αλλά όχι μόνο σε πλαίσια αποκλειστικότητας, μιλώντας όμως ε, περισσότερο για ε, περιοχές, κομοπόλεις δηλαδή, που θα μας ε, αναγάγουν σε ένα επίπεδο ανάπτυξης έτσι ώστε να μην υπάρχει αστιφιλία και απερίμωση άλλων ε, πόλεων ή αγροτικών περιοχών. Uh, I would go back Θα ήθελα να επανέλθουμε στον κύριο Κατσολίνο, αν θέλει να σχολιάσει. Όχι, δεν έχω σχόλια. Έχουμε μέχρι τον ε, Σεπτέμβριο. Θα μας απασχολήσει το θέμα τον Ιούλιο και θα συνεισφέρουμε όσο περισσότερο με Επιμένω στο εξής. Δεν υπάρχει κάποια ενωτική στρατηγική της Ευρώπης ως προς το θέμα της, των άστεων και της, και της αστιφιλίας. Μας, ενδιαφέρουν, ε, μας ενδιαφέρει ανάπτυξη του θέματος ε, στα πλαίσια, σε ενωτικά πλαίσια και όχι σε επίπεδο πόλεων μεμονωμένα. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τη νομική βάση και πολιτικές προτάσεις έτσι ώστε να προσδώσουμε στην Ευρώπη μία ενωτική διάσταση ως προς το θέμα των άστεων. Αυτή η συζήτηση είναι απόλυτα αναγκαία και αποφασιστική σημασία. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να τα εντάξουμε στην πρόταση ψηφίσματος. Η έκθεση δεν ήρθε από το Λουξεμβούργο, άρα θα έχουμε την έκθεση την, ε, το Σεπτέμβριο και θα μας πει ο κύριος Κοτσολίνο πώς εξελίσσονται τα πράγματα το Σεπτέμβριο. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα, επί το οποίο είχαμε καθυστερήσει, ίσως θα θυμόσαστε, ότι προσαρμόσαμε το νομικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έτσι ώστε να δούμε το θέμα της στέγασης της στέγασης, ιδιαίτερα των Ρωμά, και αυτό αποτελεί μία πρόκληση για τη μελλοντική μας πολιτική. Στο μεταξύ, τα κράτη-μέλη που ασχολούνται με το θέμα των Ρωμά έχουν ορίσει συνεκτικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο Γι' αυτό το θέμα της στέγασης μας απασχολεί ιδιαίτερα για την ε, ενσωμάτωση των Ρωμά στον κοινωνικό ιστό. Έχουμε για την ανταλλαγή απόψεων σήμερα μαζί μας τον Αλέξανδρο Τσολάκη, ο οποίος προέρχεται από την Γενική Διεύθυνση Ρίτζο και ασχολείται με τη διεκπαιρέωση ζητημάτων στέγασης στο ΕΤΠΑ και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας αναφέρω τι έχει συμβεί εδώ και δύο χρόνια από εγκρίθηκε η, τροποποίηση. Λίγο αργότερα ο κύριος Βανίστερ Ρόι ζήτησε από την DG Regio να δώσει κάποιο είδος σχέδιο προώθησης. Η DG Regio προτίμησε να έρθει σήμερα με κάτι που ήδη έχει γίνει και ίσως και με την αρχή μιας διαδικασίας. Όταν λάβαμε αυτό το νέο μέσο, αυτή τη νέα διευκόλυνση, Είχαμε δύο επιτακτικές ε, προσταγές. Το μία ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που προέρχονταν από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι των όσων χρειαζόταν να κάνουμε. Και το άλλο ήταν, όπως είπατε, να έχουμε να τοποθετήσουμε την στέγαση με, στο επίκεντρο των εθνικών στρατηγικών ολοκλήρωσης των Ρωμά. Ξέρω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή τη φάση, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα στοχεύαμε κάποιες χώρες ώστε να γίνει αυτή η προώθηση του άρθρου 7.2 και του μέσου. Και εδώ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Ελλάδα καθώς και η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία θεωρήσαμε πως είναι πολύ σημαντικό και η χώρα στόχος και θα επανέλθω σε αυτά. Επίσης δουλέψαμε όσο γινόταν σε διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εσωτερικό επίπεδο, δηλαδή να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε στις υπηρεσίες της Κομισιόν αυτή την, ε, αυτό το μέσο, αυτή τη διευκόλυνση, να καταλάβουν τι σήμαινε την ανάγκη για ολοκληρωμένη προσώγηση που σημαίνει και εντός της Κομισιόν συντονισμό ανάμεσα στο Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Ε, τοπικές ε, αρχές, ε, την κοινωνία των πολιτών, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που ήρθαμε σε επαφή μαζί τους έτσι ώστε να επιμείνουμε και να τους εξηγήσουμε πως αυτό το νέο μέσο θα μπορούσε να είναι ένα συγκεκριμένος τρόπος για να αποδείξουμε κάτι γιατί όταν κανείς δουλεύει ιδιαίτερα στο θέμα των Ρωμά ε, ακούει πολλές φορές ότι τίποτα δεν ε, λειτουργεί όσον αφορά την, ολοκληρω... την ένταξη των Ρωμά ιδιαίτερα για προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό πολλές φορές. Ένα μεγάλο σημαντικό τμήμα λοιπόν της στρατηγικής μας ήταν να εντοπίσουμε δήμους, κοινότητες, όπου οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών θα ήταν πρόθυμες και ικανές να εμπλακούν σε μακροχρόνια παρεμβάσεις στέγασης και με συστηματικές επισκέψεις επιτόπου για συζήτηση με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών ε, και αυτό θα ήταν ε, αναπόσταση στο τμήμα της μεθόδου εργασίας μας. Αναπτύξαμε λοιπόν συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και οι συζητήσεις που είχαμε κυρίως με τις τοπικές, την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές έδειξαν ε, σαφώς ότι η ολοκληρωμένη μέθοδος δεν μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι μια μέθοδος μεταξύ άλλων, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις ε, που όσον αφορά τη τοπική κατάσταση κάθε φορά. Τόσο πολλές διαφοροποίησεις υπάρχουν ώστε δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα συγκεκριμένο πρότυπο θα ταιριάξει για όλους. Πιστεύουμε ότι η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση ιδιαίτερα με αυτό το συμμετοχικό στοιχείο μπορεί όντως να ανταποκριθεί σε κάποιες από τις προκλήσεις. Τέλος βέβαια δουλέψαμε με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, εθνικές αρχές, που όπως ξέρετε δεν είναι πάντοτε οι πιο ανοιχτές στο θέμα της ε, ένταξης των ε, περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Θα πρέπει να πω ότι δουλέψαμε πολύ εντατικά για τέσσερις χώρες με επισκέψεις για το θέμα της ένταξης των Ρωμά και καταφέραμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο και εκεί. Τα πρώτα αποτελέσματα τώρα να σας πω ποια είναι. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τρεις ομάδες χωρών. Η πρώτη είναι η Γαλλία και η Βουλγαρία. Γαλλία-Βουλγαρία είναι η πρώτη ομάδα γιατί είναι οι μόνες χώρες όπου ήδη υπάρχουν αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας υπάρχει και μια διαδικασία για ε, ε, ε, πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις δήμους Μπουργκάς, Βιντίν, Τούρκνιτσα και Αντέρ και αυτές, αυτοί οι δήμοι έχουν επιλεγεί 10 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό ε, ταμείο Ανάπτυξης έχει, αφιερωθεί εκεί και κάποια χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο. Η διαδικασία λοιπόν που έχει ξεκινήσει ήδη στη Γαλλία δεν υπήρχε κάποια κεντρική διαδικασία με τον ίδιο τρόπο, αν και υπήρχε μια εξαιρετική εφαρμοστική εγκύκλωση για το πώς θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο 7.2 γιατί από τη μια πλευρά είχαν ε, τους ε, Ρωμά και από την άλλη τους ε, Jean de Voyage όπως τους αποκαλούν. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και εκεί τουλάχιστον 10 προγράμματα, 11 περιφέρειες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, έχουν, δώσει, έχουν λάβει 20 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής Αυτές οι δύο χώρες λοιπόν είναι οι πιο προηγμένες. Έπειτα έχουμε διάφορες χώρες όπως η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα όπου στις δύο πρώτες η πρόσκληση για υποβολή προγραμμάτων για πιλωτικές παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει, έχουν δοθεί πόροι έχουν μάλλον όχι δοθεί, έχουν ε, προβλεφθεί οι πόροι και πιθανότατα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Ελλάδα δουλεύει για ένα πολύ ενδιαφέρον πρότυπο όπου θα ε, γίνει δουλειά σε τοπικό επίπεδο με δύο πιλωτικές περιφέρειες. Η μία είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και η Θεσσαλία. και επίσης έχουν ε, ξεκινήσει την ε, κατανομή των κονδυλίων ΕΚΠΑ και ε, τροποποίηση των προγραμμάτων τους. Έχουμε έπειτα στη συνέχεια δύο χώρες, μάλλον μια πόλη και μια χώρα, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε. Η μία είναι η Όστραβα, στην Τσεχία, η πόλη, όπου είναι ο μόνος Δήμος που έχει αναλάβει πρωτοβουλία μετά από μία επίσκεψη που κάναμε. Συμφώνησε για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα καλύψει γύρω στις 6 και 8.000 με 8.000 περιθωριοποιημένους ανθρώπους, 10 γειτονιές. Έπειτα έχουν βάλει χρήματα του Δήμου για να προετοιμαστούν και θα πρέπει να πω ότι έχουν κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Δυστυχώς φαίνεται να υπάρχουν δισταγμοί από τις διαχειριστικές αρχές στην έγκριση. Κατά τον ίδιο τρόπο και στη Ρουμανία και η Ρουμανία είναι ακόμα πιο επίγουσα η κατάσταση θα έλεγα. Πετύχαμε από τέσσερις δήμους, μεγάλους δήμους, Βραήλα, Γαλάτσι, Βουκουρέστι, ένα κομμάτι του Βουκουρεστίου, το ΜΕΑΣ 2 και η Κλούς, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση με μία από τις χειρότερες καταστάσεις στην Ευρώπη όπου καταφέραμε να πείσουμε τις, ε, τους Δήμους, τις τοπικές αρχές και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την κοινωνία των πολιτών, την τοπική κοινωνία των πολιτών, τον OSI, τον UNDP, όλους να πιέσουν ώστε να ε, προωθηθούν αυτά τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Και μέχρι στιγμής παρά την επίσκεψη του Επιτρόπου που τα ανέφερε όλα αυτά, παρά επιστολή του Γενικού μας Διευθυντή. Για την ώρα υπάρχει αντίσταση. Με λυπεί πάρα πολύ αυτό και θα ήθελα να σας ζητήσω όσο μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Πάνω κάτω λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Ίσως θα μπορούσα σύντομα να σας δώσω κάποια πρώτα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει θετικά εξαιρετικά σημαντικός αντίκτυπος της ρητής στήριξης της Ένωσης για την ένταξη των Ρωμά και κυρίως για τη στέγαση. Αυτό έχει σημάνει τη διαφορά όσον αφορά την αντίληψη για το πώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο το που υιοθέτησε η Κομισιόν ε, θα μπορούσε να, να είναι ένα, μάλλον είναι ένα δυναμικό πλαίσιο με στόχο να βοηθήσει. Ε, στο τοπικό επίπεδο υπάρχει μια γνήσια συγκατανόηση και ενδιαφέρον για την ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι φυσικά παντού, αλλά όταν υπάρχει είναι γνήσιο το ενδιαφέρον και βέβαια υπάρχει και σημαντική κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών το, ε, συμπεριλαμβανομένη σε της κοινωνίας των πολιτών των Ρωμά Υπάρχει κάποια εμπειρογνωμοσύνη, αλλά η οποία είναι πολύ διασκορπισμένη και θα πρέπει να μπορέσουμε να τη συγκεντρώσουμε. Και έπειτα και παραδόξω υπάρχει και ένα δυναμικό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πίστευε κανεί πω όχι. Αλλά χρειάζεται τεχνική βοήθεια και υπάρχει εδώ πραγματικό ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνική βοήθεια και είναι πολύ πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε το τοπικό επίπεδο ώστε να μπορέσει να φτιάξει καλά σχέδια γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα. Δυσκολίες αν ε, έχουμε πάντοτε υπόψη φυσικά το θέμα των διακρίσεων και του αποκλεισμού τον Ρωμά που πάντοτε θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ως δυσχέρεια. Μια μεγάλη δυσκολία και το ξέρετε καλύτερα από μένα είναι η ασυμβατότης των διαφόρων δημοσιονομικών μέσων. για να μπορούμε να έχουμε μια ομαλή ροή στις ολοκληρωμένες αυτές τις επιχειρήσεις με την απαραίτητη ευελιξία. Αυτό έχει προκαλέσει τη τομεακή προσέγγιση στο, στις εθνικές δικήσεις, στους εθνικούς δικοτικούς μηχανισμούς και είναι κομμάτι της δυσκολίας ε, του να περάσουν αυτές οι ιδέες για ολοκληρωμένα προγράμματα δεν υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία δε στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, γιατί αυτά τα προγράμματα δεν είναι τριετή. Θα πρέπει να βγούμε από το όριο της τριετίας. Δεν θα πρέπει να καλύπτονται μόνο τα πρώτα τρία χρόνια της ε, εθνικής ε, στρατηγικής ολοκλήρωσης, αλλά και ακόμα 10-20 χρόνια μετά. Τέλος, υπάρχει ο φόβος των δημοτικών αρχών και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει στο μέλλον να το δούμε περισσότερα ε, με τον εδαφικό τρόπο ότι δηλαδή οι τοπικές αρχές κάνουν θετικά, οι δημοτικές αρχές κάνουν θετικά βήματα όσον αφορά κυρίως την στέγαση, αλλά συχνά φοβούνται να ελκύσουν ομάδες εκτός. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί μόνο να αντιμετωπιστεί όσον αφορά την δαφική συνοχή και κυρίως όσον αφορά την ε, κοινότητα το Ρωμά με δουλειά σε, σε επίπεδο υπαίθρου γιατί το 50% αυτών των χωρών, των περισσότερων χωρών, ε, μάλλον αυτών των πληθυσμών, ζουν σε περιοχές της υπαίθρου και γι' αυτό και έχουμε ζητήσει παράλληλα μαζί με το ΕΚΠΑ και το Κοινωνικό Ταμείο να ε, ληφθεί υπόψη και, η ανάπτυξη, και από το Ταμείο Ανάπτυξης Πέθρου η συγκεκριμένη κατάσταση. Τέλος, είναι προφανές ότι εφόσον η στέγαση είναι τοπικό ζήτημα, εξοχήν σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες. Πράγμα που σημαίνει ότι η προετοιμασία οποιοδήποτε προγράμματος ξεκινήσει θα πρέπει να βασίζεται στην προετοιμασία τόσο των δικαιούχων όσο και του ευρύτερου πληθυσμού ώστε να θεωρηθεί ως μια διαδικασία εξέλιξης, ανάπτυξης και όχι ως φιλανθρωπία. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψή μας για αυτά τα θέματα και να μην θεωρούμε ότι το να επενδύσουμε σε αυτή την περίπτωση στην ένταξη των Ρωμά ή στην ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων εν γέννη, ότι είναι απλά μια λύση ώστε να αποφύγουμε το πρόβλημα. Όχι. Και ως προς αυτή την έννοια θα είναι πρόκληση να δούμε πώς ακριβώς σε τοπικό επίπεδο η οικονομική δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί μέσω της κατασκευής των υποδομών και της στέγασης θα μπορέσει να ωφελήσει αυτή την ομάδα στόχο εξ αρχής ως τρόπο τοποθέτησης κάποιων από αυτή την κοινότητα στις βασικές οικονομικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Εξαιρετική η παρουσίαση και σας ε, ε, ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες που έδειξαν ότι έχετε και προσωπική πείρα επί του θάματος. Ο κύριος Λάμπερ Πανίστερόι. Ευχαριστώ εντυπωσιάστηκα από τον τίτλο εισαγωγής Implementing Housing Issues. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως με μια απόφαση η οποία έχει εγκριθεί σε σχέση με τον ε, κανονισμό για τις ομάδες τις Με, με λοιπόν αναφέρθηκε το θέμα της, ε, ε, το θέμα της κατοίκηση κτλ. Αλλά παρόλα αυτά να ευχαριστήσω τον ε, ε, κύριο, διότι αυτό ο τρόπο μας οδηγεί στο να κάνουμε και κάποιε ερωτήσεις. Ουσιαστικά τι γίνεται. Εμείς επιθυμούμε να υποστηρίξουμε μια κατάσταση η οποία είναι περίπλοκη στο κλούς. Με πλησιάσανε κάποιοι από τους ε, κατοίκους αυτού τις περιοχές από κάποια ε, ένωση με την ιδιότητα του συντονιστή προβληματιστήκαμε να δούμε αν είναι δυνατόν να στείλουμε μια αποστολή στο κλούς και πραγματικά το υποστηρίζω αυτό να πάμε εκεί να δούμε επί τόπου πώς έχει κατάσταση τι να σας πω βρισκόμαστε σε αδίέξοδο και τι θέλω να σας πω υπάρχουν άτομα που είναι μακριά από την πόλη βρίσκονται κάτω από άθλες συνθήκες θα πρέπει να είναι κανείς έτοιμος να δώσει μια νέα ευκαιρία σε αυτόν τον κόσμο. Ε, τι θα, γίνει. Ε, θα χρειαστεί ίσως, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να γίνουν νέες κατοικίες και να τους βοηθήσουμε να μπουν μέσα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πολλές φορές να πάμε επί τόπου για να έχουμε μια άμεση εμπειρία. Θεωρώ πάντως ότι είναι πολύ καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν έτοιμη, ή είναι μάλλον έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική της ολοκλήρωσης, της ένταξης μάλλον. Εγώ έχω, ε, έχω γράψει μια επιστολή στην Επιτροπή και πήρα απάντηση χωρίς να ξέρω, καταλαβαίνω τίποτα, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Αναφέρθηκε ότι ναι, ναι, ναι, θα εγκρίνουμε αυτό τον κανονισμό, Σα ευχαριστούμε λοιπά. Ξέρονται ότι 70% των πόρων που διαθέτουμε θα χρησιμοποιηθούν για αυτές τις πρωτοβουλίες, ε, αναρωτιέται κανείς πραγματικά πώς έχει κατάσταση. Στο νέο κανονισμό λοιπόν Τι γίνεται. 14-2020 έχουμε τα σωστά μέσα. Φεντέρ, Κοινωνικό Ταμείο, θα μας επιτρέψουν πραγματικά να κάνουμε κάτι καλύτερο. Μήπως χρειαζόμαστε μια πιο κεντροποιημένη, ένα κεντροποιημένο συντονισμό. Υπάρχει η ευθύνη, η τοπική Μήπως όμως πρέπει να δούμε και κάποια ε, διαδοχικά στάδια. Σίγουρα χρειάζεται μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να εντάξουμε στη διαδικασία τις τοπικές αρχές, οργανώσεις, αυτούς που αποφασίζουν, ούτω ώστε να γίνει καλύτερη χρήση των ε, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά ε, μη αποδεκτές και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τους Ρώμα. Πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε στη βάση αυτού του θέματος. Στο ΕΛΚ έχουμε λάβει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και θεωρούμε σε, στις χώρες στόχους έχουν εγκριθεί στρατηγικές, έχουν ε, καθοριστεί κάποια μέσα για την αντιμετώπιση την εφαρμογή των στρατηγικών, αλλά τα αποτελέσματα πούντα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα, έχουμε πάρει κάποιο μάθημα, ε, προβληματιζόμαστε για κάποια νέα αντιμετώπιση. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, έχουμε προβληματισμούς, ε, γίνονται, έχουμε καθίσει με το Συμβούλιο στο ίδιο τραπέζι, έχουμε διαπραγματευτεί, ε, έχουμε αποφασίσει τη διδαξή μιας έκθεση και ο, ο είναι εδώ. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, καλύτερη και σε βάθος συνεργασία. Ευχαριστώ. Thank you all. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Μπλάξεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τρέχουσα πρόταση σε σχέση με το ΕΤΠΑ, τη συμμετοχή του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να μας οδηγήσει και σε μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια τσεχική ένωση η οποία ασχολείται με θέματα και στέγασης και αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει κυρίως είναι η ενεργειακή αποταμίευση. Αυτός είναι ο πρώτος τομέας και το δεύτερο είναι η αρρωγή σε θέματα στέγασης για τις ευάλωτες αυτές ομάδες. Μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να ε, ασχοληθούμε και με ενοικίαση, διότι έχει μεγάλη σημασία η βελτίωση του πλαισίου κινητικότητας. Ίσως θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία και σε αυτούς τους τομείς, ε, δηλαδή στην ενοικίαση. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη συζήτηση αυτή διότι αποτελεί μια ακτινογραφία της τρέχουσας κατάστασης και παράλληλα δείχνει τι πρέπει να γίνει στην άμεσα επόμενη περίοδο. Επειδή προέρχομαι από τη Ρουμανία θα πρέπει να πω ότι το θέμα της στέγασης και της απόδοσης στέγασης αποτελεί μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Διότι όταν κατασκευαστούν και παραδοθούν σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, αυτό που έχει σημασία είναι η βιωσιμότητα. Πώς δηλαδή οι στεγαζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Να μπορέσουν δηλαδή να πληρώσουν το ηλεκτρικό τους, τα έξοδά τους και ούτω καθεξής. Και τι θα γίνει με τις γυτνιάζουσες περιοχές. Ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Βαλνίστερόι ότι μαζί με τον κύριο Μάτουλα πήγαμε στο Αράντ. Μεταβήκαμε στο Αράντ όπου είδατε ένα πρότυπο που μπορούμε να ακολουθήσουμε. 900 ε, Ρωμά είχαν εργασία και θα ήθελα να λάβετε υπόψη μία γερμανική επένδυση όπου μπόρεσαν σε αυτή τη γερμανική, σε αυτή τη γερμανική επιχείρηση να εργαστούν 900 Ρωμά. Έχει λοιπόν σημασία το θέμα της εκπαίδευσης, είναι πρώτης της σημασίας τη στιγμή που τα παιδιά των Ρωμά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και δεν μπορούν να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας, σίγουρα θα είναι μελλοντικοί άνεργοι. Και αυτές οι κοινότητες θα είναι υποανάπτυκτες και θα είναι πάντα εστίες εγκληματικότητας. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία, στον κοινωνικό ιστό. Το πρόβλημα είναι η εκπαίδευση. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει ένα σχήμα θετικής διάκρισης, δηλαδή από την πρώτη τάξη δημοτικού μέχρι το πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα κονδύλι για να γίνεται ε, χρήση της γλώσσας των Ρωμά και έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μπορούν να κλείσουν τον κύκλο σπουδών γιατί προβλέπεται και η γλώσσα των Ρωμά. Θα ήθελα να πω λοιπόν στον κύριο Τσολάκη ότι έχει μεγάλη σημασία να ε, λάβουμε υπόψη την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στην επιλεξιμότητα των σχεδίων προς χρηματοδότηση. Δηλαδή, ως προς το Ταμείο της Συνοχής και το ΕΤΠΑ, καθώς και τα κοινωνικά ταμεία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι το 2014. Να δούμε δηλαδή τι θα γίνει μέχρι το 2014, διότι αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση τώρα και περιμένουμε μέχρι το 2014, θα επιταχυνθεί το πρόβλημα των Ρωμά. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτές οι κοινότητες να κινηθούν προς τον πολιτισμό προς τις ε, κοινωνίες, την κοινωνία του 21ου αιώνα. Εάν δεν ε, δημιουργήσουμε ελίτ και σε αυτές τις κοινότητες, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ούτω καθεξής, για να βοηθήσουμε αυτούς τους φορείς, εάν δεν δημιουργήσουμε αυτές τις ελίτ που θα δημιουργήσουν πρότυπα και σε επίπεδο Ρωμά, τότε δεν θα φτάσουμε πουθενά. Θα πρέπει να προωθήσουμε τους δικούς τους ηγέτες και όχι να προβάλλουμε ηγετικά πρότυπα απ' έξω. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις τοπικές ελίτ των Ρωμά. Έτσι ώστε να ξεφύγουμε από κλισέ να ξεφύγουμε από ρατσιστικά πρότυπα, τα οποία βλέπουμε και σε δημοκρατικές ε, κοινωνίες. Εάν δεν ξεπεράσουμε όλα αυτά και δεν έχουμε έναν επιχειρησιακό διάλογο, τότε δεν θα φτάσουμε πουθενά γιατί πολλές φορές οι ελίτ έχουν και προσωπικά συμφέροντα. Εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε ελίτ οι οποίες θα απελευθερώσουν τις κοινότητες των Ρωμά. Μόνο μία ευρωπαϊκή απάντηση θα μπορούσε να δοθεί στο θέμα των Ρωμά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας υπενθυμίζω το θέμα κατοικία είναι ένα μεγάλο δικαίωμα το οποίο είναι γραμμένο στα, στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και όντως σήμερα όταν βλέπουμε τις στατιστικές και κυρίως τις άσχημες συνθήκες στην κοινότητα το Ρώμα, βλέπουμε ότι πλήττονται κυρίως τα παιδιά. Μιλάμε για άσχημες συνθήκες λοιπόν κατοικίες και πραγματικά αυτό έχει επιπτώσει και στην υγεία θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από το 11 στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ έχουμε αυτό το μέσον και είναι το μέγιστο που έχουμε στα χέρια μας. Εμείς στη Γαλλία έχουμε πολλά προβλήματα. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές που έχουν διαγράψει το στόχο τους λαμβάνοντας υπόψη και το κλίμα Το θέμα είναι αν αυτό το ποσοστό που έχουμε στη διάθεσή μας ε, στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ αρκεί για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ορισμένες κοινότητες χρησιμοποιούν αυτά τα, αυτούς τους σπόρους, τα κονδύλια, για, ε, όχι για την κατήγηση, αλλά για υποδοχή. Τους επιτρέπει το γαλλικό κράτος να δράσουν έξι. Βλέπουμε δηλαδή από μία χώρα στην άλλη η νομοθεσία είναι διαφορετική, άρα μπορεί να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Τώρα έχουμε το στόχο 2014-2020. Η Γαλλία στοχεύει, θέλει να εξασφαλίσει, να εγγυηθεί περισσότερη συνέργεια που λέμε ε, του ΕΦΣΕ και του ΦΕΝΤΕΡ, διότι όπως το είπατε αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της καρκίσης είναι το σημαντικό, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία βρίσκονται σε σχέση, ε, είναι παρεμφερή σε σχέση με αυτό το θέμα. Εγώ σκέφτομαι το σύνολο των δημοσίων ε, υπηρεσιών. Ε, ε, οι πληθυσμοί αυτοί πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, τρεχούμενο νερό. Αυτό που λείπει σήμερα είναι μια πραγματική αληθινή πλατφόρμα η οποία να δείχνει και να συνεργάζεται, να μάλλον να εκμεταλλεύεται και την εμπειρία των διαφορετικών κοινοτήτων. Υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες. Υπάρχουν συνεργασίες, αλλά πολλές φορές ε, έχουμε κοινότητε οι οποίες δεν έχουν καμιά ιδέα για αυτή την εμπειρία. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή την εμπειρία και να υπάρξει ένα σχέδιο πιο γενικό, πιο ολοκληρωμένο. Επίσης να δώσω μια έμφαση ότι ε, το θέμα της κατοικία είναι ας πούμε ε, η πηξίδα, ο άξονα πάνω στο οποίο κινούμαστε. Αλλά να γίνει κατανοητό Υπάρχουν πάλι περιοχές, σε διάφορες περιοχές έχουμε ε, ε, κατοικίες οι οποίες είναι ε, άδειε, εγκαταλελειμμένες, που δεν τις εκμεταλλεύεται κανείς. Θα μπορούσε κανείς να τις χρησιμοποιήσει πραγματικά στη συγκεκριμένη περίπτωση ή δυνατόν για τους Ρώμα. Ευχαριστώ. Πρέπει να ψηφίσουμε στις 10 και 4 και έχουμε ακόμα δύο ομιλητές. Η κυρία Σιριγκόγιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που άφησαν το θέμα οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα να ε, σας συγχαρώ και να μας συγχαρώ, γιατί εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του ΕΤΠΑ για τους Ρωμά. Αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε από, ότι από την εποχή του Φελίπε Γκονθάλεθ ε, καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης ε, και συνύπαρξης των Ρωμά. Και έτσι είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων και σχέσεων μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού ιστού. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να προωθήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές υπέρ των Ρωμά και έχει σημασία να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ κοντά μας η Ρωμά, γι' αυτό θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, να τους εντάξουμε στον εκπαιδευτικό ιστό. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την επιτυχία των προγραμμάτων μέσα στα πλαίσια του ΕΤΠΑ και τη συμμετοχή ε, της γραμματείας των Ρωμά. Και είναι γεγονός ότι συμφωνώ με τον ε, κύριο Τσολάκη ότι χρειάζονται ε, συγκεκριμένα προγράμματα για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε πλήρως. Ο κύριος Μάτουλα. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος και να μην ε, επαναλάβω τα όσα προαναφέρθηκαν διότι ο συνάδελφος Μποστινάρου έθιξε ένα θέμα ουσίας ως προς την προσέγγιση. Ε, είχαμε μία μελέτη, έγινε και μία επίσκεψη στο Αράντ σε ένα οικισμό όπου κατοικούν χίλιοι Ρωμά και όπου συμμετέχουν στον ε, εργασιακό ιστό. Δεν κάνουμε λάθος εμείς ως Ευρωπαίοι όταν πάντα φύγουμε το θέμα των Ρωμά γενικά χωρίς να το δούμε αναπερίπτωση. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα μίας ποσοστιαίας αναλογίας μέσα στην όλη κοινότητα των ορμά. Εάν μιλάμε για το πρόβλημα των κοινοτήτων των Ρωμά, αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε και τα αποτελέσματα στα οποία φτάνουμε, αυτά αποτελέσματα, γιατί επανερχόμενος αυτούς τους ενταγμένους Ρωμά, Εκείνοι δεν θέλουν ε, να γίνεται λόγος για προβλήματα της κοινότητας των Ρωμά, διότι έχουν ενσωματωθεί και δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Ενώ εμείς πολύ συχνά μιλάμε για τους Ρωμά γενικά. Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με τα κονδύλια για τη στέγασή τους. Ο κύριος Σολάκης στην παρουσίασή του μίλησε για το πρόβλημα της ασυμβατότητας ορισμένων χρηματοδοτικών μέσων. Δηλαδή πολλές φορές το ότι δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση ή εγγραφή πιστώσεων για σχέδια στέγασης εμείς στη Ρουμανία έχουμε σχέδια ενσωμάτωσης μέσω κοινοτικών προϋπολογισμών, προϋπολογισμών δηλαδή προϋπολογισμών των κοινοτήτων όπου εγγράφονται και ενσωματώνονται κοινωνικά κονδύλια. Γι' αυτό θα πρέπει να πλουστεύσουμε αυτό το μηχανισμό χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων εάν θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Διαφορετικά θα μείνουμε στο ίδιο στάδιο, δεν θα γίνει σωστή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και θα υπάρχουν ε, μεγάλες δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες και έχω να σας δώσω αυτά παραδείγματα. Οι συνάδελφοι επισκέφθηκαν συγκεκριμένους οικισμούς, εκατοντάδες οικισμούς που χρηματοδοτήθηκαν από τις τοπικές κοινότητες και όχι από κοινοτικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν απορροφώνται εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος ε, Τσολάκης θα ήθελε να σχολιάσει. Δεν είναι ανάγκη να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, διότι δεν εντάσσονται στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλώς θα σταθώ σε ένα σημείο τη στέγαση. Η στέγαση είναι λύση. Δεν είναι η λύση, αλλά μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα εάν δεν έχει προγραμματιστεί σωστά και έχουμε πληθώρα παραδειγμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε καλή προετοιμασία αυτών των σχεδίων και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει βάθος χρόνου έτσι ώστε να μπορεί να φτάσει σε βιώσιμα σχέδια και για να μπορέσει να εντάξει όλες τις δυνατότητες υποστήριξης μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση. Νομίζω ότι με βάση αυτή τη συζήτηση και τα θέματα που θίγησαν θα πρέπει να δούμε το θέμα της γενικότερης πρόκλησης δηλαδή στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι διατάξεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε με αυτή την ε, μεγάλη πρόκληση της ένταξης των Ρωμά και να έχουμε αυτή την εσωματωμένη προσέγγιση έτσι ώστε και στις αστικές περιοχές και στις αγροτικές να υπάρχει μια σοβαρή προσέγγιση. Το δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο με βάση αυτές τις ε, συζητήσεις θα ήταν σκόπιμο να υποβάλω μια επιστολή στον Επίτροπο Χάν έτσι ώστε κατά τη διαπραγμάτευση οικονομικών εταιρικών συμφωνιών, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα και το αναγνωρίζουμε, το θέμα αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι για τη βελτίωση της κατάστασης, ε, αν όχι για την επίλυσή της. Εάν δεν αντιτίθεται κάποιος, θα αποστείλω αυτή την επιστολή. Ωραία, θα αποστείλω την επιστολή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση και συμμετοχή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία πρέπει να ελέγξουμε τα μηχανήματα, γι' αυτό βάλτε τις κάρτες σας για να γίνει η δοκιμή. The check. We will ask Miguel to open the vote. So we are opening the vote. Αρχίζει η ψηφοφορία. Miguel. Yes. It's not opened. No. Not working. Well, So what? Ωραία, θα μας ενημερώνετε. Εάν δεν συμβαδίζετε με το ΕΛΚ θα μας ενημερώνετε γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Μπορείτε να ζητήσετε από το βοηθό σας να σας φέρει την κάρτα σας. Ψηφίσατε όλοι, δοκιμή. Oh, it's moving, so I don't know whether you are not yet ready or... Okay, we close the... πέρας. Ωραία. Σημείο 10. Η έκθεση της ε, Μαρία Ριγκόιαν Πέρες. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Διακόπτη πρόεδρος. Once again, sorry. Amendment 77. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν σας βλέπω καλά, γι' αυτό όταν σας ζητάω να σηκώσετε το χέρι σας να το κάνετε ευκρινώς. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ε, συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 95 υπέρ κατά πάλι 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ Κατά. Θα ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 110. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός, λέει η πρόεδρος και διακόπτη. Ναι, εντάξει, και εσείς είσαστε υπέρ. Επτά, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. 125 αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται, νομίζω. Ωραία, σε ελέγξουμε. 134 αρχίζει η ψηφοφορία. vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται, απορρίπτεται πράγματι. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 150. Αν θέλετε να ελέγξουμε, εντάξει. 149 ελέγχουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σημειώσμος 13 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβασμός 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. Όχι. Απορρίφθηκε άρα δεν καταπίπτει. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά ελέγχουμε. 176 έλεγχος. Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται πράγματι. 177 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 17 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 καταπίπτει όχι, όχι, ψηφίζουμε, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 230... Όχι, όχι, 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. «236» νομίζω λέει πρόεδρος διότι καταπίπτει η 230, η 235, έτσι δεν είναι. So tell me what, what I should vote, and, and it's just the result. 236. So as I said, 200... Ωραία, ψηφίσουμε 236 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 237 παρόμοιες, παρόμοιες, πανομοιότυπες. Ωραία, ψήφισαμε και τις δύο. Συμβασμός 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 55 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. 256 ελέγχουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. closed. And it is απορρίπτεται. 257 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 263 τι θέλετε, 263 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβασμός 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 30 και 267 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 270 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 271 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 272 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 274 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σύμβασμος 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μεγάλος αυτός ο συμβιβασμός δεν λέει να τελειώσει Ωραία. Αυτό, αυτό θα πει συμβιβασμός. Αυτό θα πει συμβιβασμός. Τετρασέλιδος, αιτιολογικές σκέψεις, 28 ε, υπέρ κατά από, ε, εγκρίνεται. Α, όχι έκανα λάθος. τι έκανα, τι έκανα λέει η πρόεδρο. 37, 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά ας ελέγξουμε ελέγχουμε παρακαλώ για την 66 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρασα. δεν ψηφίσατε όλοι εγκρίνεται η 66 ήταν αυτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. We close. Πέρας. Δεν ψηφίσατε όλοι, αλλά πρέπει να κλείσουμε 36 προς 1 και 6 αποχές. Συγχαρητήρια. Δεν ήταν εύκολο να σας συγχαρούμε. So... We go to point 11 on our agenda, which is... Σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη ψηφίζουμε την έκθεση Αλφονσίν, μακροοικονομική, μακροπεριφερειακή στρατηγική. Easier vote, I hope. Okay. So we go to amendment 23. Who is in favor? Who is against? Abstentions adopted. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Abstentions adopted. 28 in favor. 28 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ. Μου είπα ότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ότι πρέπει να μπει στο υπάρχον κείμενο και λέει να προσφέρει ένα πρόγραμμα δράσης και όχι ένα, μια κοινή προοπτική. Οπότε μου είπαν υπάρχει συμφωνία γι' αυτό. Αν όντω σημαίνει αυτό, να προτείνω αυτό το, την αλλαγή του κειμένου. Κοινό πρόγραμμα δράσης αντί για κοινή προοπτική. Α, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι κανείς κατά, οπότε ψηφίζουμε. Συμβιβαστική 4. Με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52. Υπέρ κατά να ελέγξουμε την 52. Ψηφίζουμε. We close the vote. Τέλος της και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά απο... ελέγχουμε την 68 ψηφίζουμε παρακαλώ τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 69 υπέρ κατά και τώρα ελέγχουμε την 69 Εγκρίνεται 24 προς 19. 74 υπέρ, ε, συγγνώμη, 70 υπέρ κατά αποχές, ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ κατά Α, δεν ξέρω. Ελέγχουμε την 72. We close the vote. And it's 25 to 20 adopted. A compromise. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 82 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 82 παρακαλώ τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 28 υπέρ 16 κατά Περνάμε στα εκτιμώντα τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στα εκτιμώ, στις ετουλικές σκέψεις 5, συμβαστική 12, υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται, συμβαστική 13, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, τροπολογία 11, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές νομίζω πως εγκρίνεται κανείς δεν θέλει έλεγχο 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Τμήμα 1 του 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα 2 της 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τμήμα 1 της 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 τους 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Περνάμε στο σημείο 12, Αλέν Καντέκ. στρατηγική για την περιοχή του Ευρωπαϊκού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τροπολογία, 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. 11 έχουμε μία προφορική, είναι κάποιο. αντιτίθεται κάποιο, όχι, ψηφίζουμε. 11 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός, όχι με συγχωρείτε, 15 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω θα ελέγξουμε τη 15. The vote is closed and it is 23 to 20 so it's adopted. 16 in favor. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, δεν ξέρω, ελέγχουμε την 33. We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 Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Συμβασμό 7. Το ξέχασα. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Βλέπετε εγκρίθηκε. 43. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε και πάλι. 43. Αρχίζει η ψηφοφορία. vote is open. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47, με συγχωρείτε συμβασμός 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 και 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός όχι 69 60. όχι με συγχωρείτε συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τις υποδείξεις Επιτροπής Μεταφορών και Μεταφορών. Τραν. Ε, ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές, πάλι πάλι λέει η πρόεδρος, για την 8, 8 υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται. Έχετε μου εμπιστοσύνη, τελική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Πέρας 39 υπέρ συγχαρητήρια. Τώρα περνάμε, πηγαίνουμε για τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Συμβασμός 1 υπέρ. Έχει εγκριθεί. We go to amendment 5, right? Who's in favor? Who's against? Abstentions, it's adopted. Εγκρίθηκε. Προχωράμε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολο... 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβασμό Αντροπολογία 19 υπέρ, αποχές εγκρίθηκε. Για την 20 έχουμε συγχωριστή ψηφοφορία. Για το πρώτο μέρο υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Για το 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμό 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμό 7 υπέρ, αποχές κατά εγκρίθηκε. Συμβασμό 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ, κατά, να το εγκρίνουμε ηλεκτρονικά, να το επαληθεύσουμε συγγνώμη ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχει εγκριθεί λοιπόν. Τώρα, στην 28 πάμε, δεν κάνω λάθος. Υπέρ για την 28 τώρα, κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 με προφορική τροπολογία δεν υπάρχει, κατά, δεν υπάρχει κάποιος που εναντιώνεται υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 Έχουμε χωριστεί ψηφοφορία πρώτο μέρο υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο μέρο έχει αποσυρθεί. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 ε, υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίθηκε. 44 υπέρ, κατά. Για να κάνουμε μια απελήφθηση ηλεκτρονικά για τι 44 παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορία. Έχει εγκριθεί με πολύ... 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρουμε. Για να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Ε, έχει εγκριθεί. Τέλος. Ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Δεν, έχει ψηφίσει, δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Ε, 39, μεγάλη, ευρία πλειοψηφία, συγχαρητήρια. Τώρα πάμε στο σημείο 14, Γιάννης Γκέιερ, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είσαστε έτοιμοι. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. 8. Ε, καταπίπτει. Περνάμε 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9, 51, 52 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκριθήκαν. 53 υπέρ, κατά αποχή απορρίφθηκε. Συμβιβασμό 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία για την παράγραφο 4, παράγραφο 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 13, 59, 60 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68-69 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 17-20-71 κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνθηκαν. 72 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 73 υπέρ κατά αποχές. Οπ. Είσαστε κατά εσείς κύριε άρα εγκρίθηκε, εντάξει. Ε, 75, χωριστή πληροφορία, ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίφθηκε δυστυχώς, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 και 74 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται, 76 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 1977-78 από κοινού υπέρ κατά αποχές εκριθήκαν 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 80 επίρ κατά αποχές απορρίφθηκε 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία για το άρθρο 9 παραγραφό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 86 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία για το άρθρο 12 παραγραφό υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 89 υπέρ κατά. Για να το δούμε ηλεκτρονικά. Για την 89 πρόκειται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Έχει εγκριθεί λοιπόν. 22 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ. Κατά. η ε, ηλεκτρονικά την 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Έχει απορριφθεί. 91 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. 92 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. Προχωρική για το άρθρο 20 παράγραφος 2α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90, 23 υπέρ. Να, συγγνώμη, 23, 93 από κοινού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Ε, Αιτιολογική σκέψη. 24. Ε, υπέρ, κατά. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Έχει απορριφθεί. 1, 25, 26 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν. Πάμε στο 2.28.29 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκαν. Συμβασμός 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Λοιπόν, 4.35.36 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 5.38.39 υπέρ, πιο, κατά αποχές εγκριθήκαν. 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκαν. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκριθήκαν 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 6-43-44 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 7, 45 και 46 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Και τώρα η τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 38 υπέρ. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Πολύ καλά. Και τώρα πάμε στην Μόιτσα Κλέβα. Έχουμε μια γνωμοδότηση εδώ πέρα για τα καινοτόμα χρηματοσυστικά μέσα στο πλαίσιο τη επόμενη πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Έτοιμη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ. Την έξι να τη δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία και έχει απορριφθεί. 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε για την 9 τροπολογία υπέρ, κατά. Νομίζω ότι απορριφθήκε, για να το δούμε, Ελίζαμπεθ. Για την 9 πρόκειται. Άρχεται η ψηφορία. Όλοι ψηφίσανε. Έχει απορριφθεί, έχει απορριφθεί. 10 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, ε, νομίζω εγκρίθηκε. 14 υπέρ, κατά. Τι έγινε. Όλοι νομίζουν ότι απορρίφθηκε. Περνάμε στις 16. Θέλω να τα επαληθεύω τα πράγματα. Καλύτερα να το επαληθεύσουμε. Έτσι μου αρέσει. Ε, ε, για τη 14 πρόκειται. Για να δούμε. Ε, όντως, λέει, απορρίφθηκε. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ Κατά. Ξανά, δεν είμαι σίγουρη. Για να, ε, συγγνώμη, να το παλιδεύσουμε ηλεκτρονικά. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Και όντω απορρίφθηκε. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίθηκε. Και ψηφίζουμε για την τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Καλώς. Τα πάμε καλά με την ώρα. Λοιπόν, αποτέλεσμα ευρεία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Dear colleagues, if you, uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώσαμε τις ψηφοφορίες πιο νωρίτερα και το τελευταίο σημείο ήταν για τις 11.30. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η Κομισιόν όμως λείπει. Όχι, κάποιος είναι, κάποιος έχει έρθει από την Κομισιόν we can, uh, he will be coming, so we can I, I don't, ask the rapporteurs if they want to... Colleagues, it all it's in the hands of the rapporteurs, I don't know where... To... Οι εισηγητές θα μας πούν ε, πού είναι ο Λαμπέρ, να αρχίσουμε τώρα ή να διακόψουμε. Αρχίζουμε. Yeah. Δεν έχουμε εκπρόσωπο από την Κομισιόν. Dear colleagues, is everybody να αρχίσουμε τη συζήτηση τώρα για τον, ε, τις κοινέ ε, διατάξεις του κανονισμού ή να το δούμε σε μισή ώρα. Uh, can Κατάλογος ομιλητών, παρακαλώ. Γιατί αν το αναβάλουμε και κανένας μετά δεν θέλει να μιλήσει, τι θα γίνει afterwards. Λαμπέρ uh, και Κωνσταντς. Ο κύριος Λούχαν λέει να αναβάλουμε τη συζήτηση κατά μισή ώρα. Βανίστελ Ρόι πολλά μέλη είναι εδώ. Ή μόλις ψηφίσαμε, θέλουμε να ε, ακούσουμε τους άλλους συναδέλφους γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις τροπολογίες. Γι' αυτό ίσως έχουμε τώρα τη δυνατότητα. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Άρα συνεχίζουμε τη συζήτηση. Θα θέλαμε τα σχόλια σας και ο Ιαν θέλει κάτι να πει. I just used the possibility that Lambert will comment my uh, intervention. Ο Ιαν Όλμπριχτ. Ας καθίσουν και οι βοηθοί. Συζητούμε το θέμα 16. Ο Γιάν Όλμπριχτ έχει το λόγο. Χτες αρχίσαμε τη συζήτηση για τις ε, τροπολογίες του κοινού κανονισμού, του γενικού κανονισμού και είναι αλληλένδετοι αυτοί οι κανονισμοί. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί ορισμένες αποφάσεις άπτονται και σχετίζονται με τους επόμενους κανονισμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε ότι ως Επιτροπή θέλουμε μία ε, κοινή προσέγγιση σε αυτούς τους κανονισμούς. Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στο γενικό κανονισμό που θα έχουν επιπτώσεις ε, στα πλαίσια του ΕΤΠΑ και ούτω καθεξής. Καταρχήν έχουμε τη συζήτηση ε, μεταξύ και κοινωνικού ταμείου. Άρα είτε θα έχουμε ένα σαφές ποσό για το έτπα και το κοινωνικό ή θα έχουμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, μετά έχουμε τους θεματικούς στόχους Δηλαδή είναι οι περίφημοι 11 στόχοι και αποτελούν το πλαίσιο για τον επόμενο κανονισμό. Γι' αυτό μιλάμε για τους θεματικούς και στον επόμενο κανονισμό θα έχουμε τα όρια. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία πώς θα αντιμετωπίσουμε τους θεματικούς στόχους και νομίζω ότι οι εισηγητές ε, έχουν ε, μία σαφέστατη αντιμετώπιση. Το τρίτο στοιχείο είναι το μέσο ε, Connecting Europe. Το συζητήσαμε χτες. Είχαμε μία ειδική έκθεση, ένα γενικό έγγραφο, αλλά εγώ πρότεινα διάφορες αλλαγές και τροπολογίες σε σχέση με το μέσο Connecting Europe γιατί όπως σας είπα έχει άμεση σχέση με την πολιτική συνοχής. Γι' αυτό και έχουμε την πρόταση διαγραφής του Connecting Europe. Και οι υπουργοί στο Βουκουρέστι ζήτησαν να αλλάξει η θέση του Connecting Europe από το 1B στο 1A, δηλαδή πέρασε από την πολιτική συνοχής στις μεταφορές και την ανάπτυξη. Γι' αυτό σας εξηγώ και τις τροπολογίες. Επίσης, μας ενδιαφέρει και το κοινωνικό, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν ξέρουμε τι, γιατί έγγραφο θα πρόκειται. Αυτό που έχει σημασία είναι να μας πούν οι εισηγητές ποια είναι η θέση τους ε, ποια είναι η θέση τους για τις εταιρικές συμβάσεις διότι οι διαρθρωτικές εταιρικές συμβάσεις άπτονται των κανονισμών. Τι θα γίνει μετά τις τροπολογίες για τις εταιρικές συμβάσεις. Εδώ ε, ε, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, διότι δεν έχει τελειώσει ο χρηματοοικονομικός κανονισμός. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε στον γενικό κανονισμό, διότι είναι η βάση για όλους τους κανονισμούς και αν ε, συμφωνήσουμε στους συμβιβασμούς, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτός τους συγκεκριμένους συμβιβασμός. Γι' αυτό έχει σημασία τι κατευθυντήριες γραμμές, ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Απλώς ήθελα να υπογραμμίσω και να πω ότι θα πρέπει να δούμε αυτό το μεγάλο μοχλό και όγκο τροπολογιών και αυτό δεν αμφισβητεί την προσέγγιση η οποία, την, προσέγγιση την οποία προωθούμε. Όσον αφορά τις δικές, μας, τις δικές μου προτάσεις, είδα στη συνέχεια ότι πολλές από τις τροπολογίες μου εντάσσονται στις προτάσεις που οι ίδιοι οι συγητές ενέταξαν για την αλλαγή του κειμένου της Κομισιόν. Ε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη σύμπνοια και έτσι θα μειωθεί ο όγκος των τροπολογιών που μας οδηγεί σε σοβαρές σκέψεις. Επειδή έχω παρέμβει τους περισσότερους, τους ε, προηγούμενους μήνες μαζί με τους συνεισηγητές, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει οικονομική μακροαιρεσιμότητα στον προγραμματισμό και στην απόδοση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Μιλάμε για ένα αποτελεσματικό απόθεμα το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μία βελτίωση του προγραμματισμού. Και από την άλλη πλευρά κυρώσεις. Αυτά εντάχθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής και ανέρεσαν εν μέρη τον στόχο βελτίωσης. Και γι' αυτό δέχτηκαν τις τροπολογίες μου οι εισηγητές. Μιλάμε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο των τοπικών φορέων μέσα στα πλαίσια των εταιρικών συμβάσεων και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού να μας υποστηρίξει γιατί μέσα στα πλαίσια της ίδιας της Επιτροπής Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το περιφερειακό επίπεδο. Μιλάμε για μία συμφωνία η οποία θα φτάσει στον απότερο στόχο της. το κοινό στρατηγικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε κατεξιοδότηση πράξη. Θα πρέπει να έχει το βάρος μιας νομοθετικής πράξης. Γι' αυτό υπέβαλα μια τροπολογία η οποία θα πρέπει να τύχει της υποστήριξης των άλλων συναδέλφων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι άλλο για μένα σημαντικό. Αυτή τη δύσκολη στιγμή μπορώ να κατανοήσω το ότι υπάρχει μία μικρή εκτροπή, αλλά δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε και για την προώθηση όλων των ε, πολιτισμικών παραμέτρων. Γιατί αυτή η έλλειψη θα σήμαινε λανθασμένη στάση των χωρών. Σημαίνει ότι απομακρύνουμε τον πολιτισμό τη στιγμή της κρίσης. Γι' αυτό θα πρέπει το θέμα αυτό να είναι στρατηγική σημασίας. Το δεύτερο θέμα αφορά την αστική ατζέντα. Μας ενδιαφέρουν οι παρεμβάσεις των παρελθόντων μηνών και η θέση μας κατά την έγκριση διαφόρων εγγράφων μέσα στα πλαίσια της αστικής ατζέντα. Χαίρομαι λοιπόν διότι έχουμε να κάνουμε με μία σύγκληση από πολλούς συναδέλφους. Εν κατακλείδη, ελπίζω αυτή η στάση σύγκληση στην Επιτροπή να αποτελέσει όθηση για να δείξουμε μεγαλύτερο άνοιγμα προς, ε, να υπάρξει μεγαλύτερο άνοιγμα προς εμάς. Καταρχήν, θα ήθελα να υπογραμμίσω την πολύ καλή εργασία των εισηγητών. Ζητήσαμε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις θεματικές ενότητες γιατί θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και στις ποσοστιαίες αναλογίες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περιφέρειες που εντάσσονται για πρώτη φορά και γι' αυτό θα πρέπει να απαλληφθεί το 5%. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε 5% βελτίωση. Επίσης, θέλαμε να ληφθούν υπόψη οι χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης για να δούμε πώς ε, έχει και πώς εξελίσσεται ο κανονισμός. Να δούμε την πραγματικότητα της ε, κάθε χώρας, γιατί η κατάσταση του 2008 δεν είναι η ίδια με την τωρινή. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε δείκτες για τη γύρανση του πληθυσμού και σε σχέση με την ανεργία, την απασχόληση, και είπαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές με νησιωτικό χαρακτήρα. Like Κάποιος άλλος θέλει το λόγο? Εάν όχι, θα θέλαμε οι εισηγητές να ασχοληθούν ή να, να σχολιάσουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι λίγο είμαι εκτός. Ε, έχω χάσει λίγο τα νερά μου. Τέλος πάντων. Ας μιλήσουμε σοβαρά. Γίνανε ε, παρατηρήσεις από τον εισηγητή και από τη σκιώδη εισηγήτρια που με πείθουν ότι πρέπει να τηρήσουμε τις μεγάλες μας κατευθυντήρες γραμμές και έχουμε εδώ με το παράρτημα του νομικού παρατήματος θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες αλλά αυτό που πρέπει να δούμε ένα σύνολο να το δούμε σφαιρικά και ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχει κανείς την εντύπωση ότι δεν ε, γίνεται κατανοητό τι έχει γίνει από την Κομισιόν ούτε από τη δική μας Επιτροπή όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Ε, βρισκόμαστε σε ένα, ε, ε, όμως σε ένα στάδιο που δεν μπορούμε να πάμε προς τα πίσω. Όπως ελέγχθηκε χθε, το θέμα είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το μέσο για να πετύχουμε ε, μια ευελιξία. Ε, αλλά θα ήθελα να πω ότι καταρχήν ότι είναι ένα από τα αποτελέσματα τα πιο σημαντικά που έχουμε πετύχει με την ε, έμφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να επιμείνουμε να την υποστηρίξουμε αυτή τη θέση έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση στην επιρροή που μπορούμε να έχουμε. Να μην περιμένουμε δηλαδή θα γιάνει η άλλη πλευρά. Τώρα, ελέγχθησαν πολλά σε γενικές γραμμές. Η ευελιξία είναι πολύ σημαντική, όντως. Αλλά θεματικά θα πρέπει να δώσουμε μια έμφαση που είναι ένα από τα σπάνια σημεία για αυτή την πολιτική. για μια σύγχρονη, εξυγχρονισμένη πολιτική συνοχή. Εδώ δηλαδή για να πετύχουμε αυτό το στόχο μας πρέπει να έχουμε δώσουμε έμφαση στη θεματική προσέγγιση. Στον Γιάννε θα έλεγα ότι δεν είναι δηλαδή πρόβλημα το να έχετε μια, ένα μεγάλη γκάμα επιλογών δεν εμποδίζει αυτό να έχει κανείς μια, ε, έτσι, ένα, μια συγκέντρωση, μια έμφαση θεματική. Η έγκριση αυτού του κανονισμού είναι το πιο σημαντικό πράγμα για, τις επόμενες, για τα επόμενα χρόνια. Από τότε ψηφίσαμε για το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο. Καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα διακυβευόμενα και ισχύει αυτό και για το θέμα, για την πρόταση που γίνεται για το ΦΕΝΤΕΡ, κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλουμε να υπάρχει κάποια εξαίρεση όσον αφορά τη θεματική προσέγγιση. Θέλουμε να υπάρχουν πιο ευρείες δυνατότητες επιλογών. θέλουμε ξανά να δώσουμε μια έμφαση να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το ότι δίνουμε έμφαση και ενίσχυση στην οικονομία και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την περιφερειακή πολιτική. Ε, επίσης υπάρχει πτυχή που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Στη Βεσφαλία, στη Βόρεια Ρινανία. Είναι σημαντικό να δεις τι κάνει αυτή η περιοχή. Δηλαδή το ότι προχωράει, προσαρμόζεται στις ανάγκες της. Και ότι έχει υιοθετήσει την τεχνολογία της πληροφορίας έχει βοηθήσει διάφορε δραστηριότητε. Αυτούς που κάνουν ποδήλατο, Φέρπιν. Ένα τουρισμός σε σχέση με αυτούς που αγαπούν να κάνουν το ποδήλατο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και ενισχύουν την οικονομία, δημιουργούν ανάπτυξη και βοηθούν την οικονομία να βγει από την παρακμία. Το πώ θα γίνουν όλα αυτά φυσικά είναι ένα μέρος που έχει ε, μια πτυχή που αφορά τι λεπτομέρειε αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τους στόχους μας. Να δούμε γενικά τι θέλουμε να πετύχουμε και μετά να δούμε τις ιδιαιτερότητες και τους κανονισμούς που πρέπει να ισχύουν. Τώρα, Connecting Europe. Εδώ υπάρχει μια σπασοκεφαλιά θα έλεγα. Μπορεί κανείς να το καταλάβει κανείς σαν ένα μέτρο το οποίο λίγο το πάει πολύ μακριά. Αυτό μπορεί να είναι μία άποψη εγώ δεν ξέρω αν εσείς καταφαίνετε και ζείτε με, με αγάπη και, και δροσερό αέρα, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια, κάτω από ποιο τίτλο. Σαν ε, εισηγητές εμείς είπαμε με αυστηρότητα ότι δεν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε ένα κεντροποιημένο τρόπο διαχείρισης αυτού του προϋπολογισμού. Θέλουμε επίσης να συνεργαστούμε για την τρόπο με τον οποίο θα γίνει η χρήση, η εκτέλεση αυτών των κονδυλίων. Ε, θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά μάλλον ίσως καλύτερα να σταματήσω εδώ. υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Θα επανέλθω. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεστε εσείς, αλλά θα επανέλθω σίγουρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Κωνσταντς. Εντάξει, αν ε, πρέπει να είμαστε σύντομοι, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ίσως μόνο κάποιο σχόλιο σε σχέση με τα όσα είπε ο Γιάνν. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι τροπολογίες θα τροποποιηθούν ε, σύμφωνα με τον κανονισμό και το περιεχόμενό του. Αλλά νομίζω πως έχουμε ήδη πολύ παράλληλη δουλειά να κάνουμε, πράγματα τα οποία ήδη έχουν προσαρμοστεί και πρέπει να προσέξουμε τις αντιφάσεις Νομίζω πως ο γενικός κανονισμός ε, είναι σφαιρικός εδώ. και για μας δεν υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα. Ίσως κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα πρέπει ακόμα να ρυθμίσουμε. Και όσον αφορά την ε, Επιτροπή Απασχόλησης, πιστεύω πως ούτε εκεί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Θα το δούμε αυτό. Äh, ich habe das ja gestern schon betont. in richtig,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 έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ναι μεν έναν ε, βασικό κανονισμό, αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς νομική βάση. Ε, ξεπερνά τον, ε, τα συνηθισμένα μπορούμε να λάβουμε υπόψη την ε, μακροπεριφερειακή στρατηγική και να την ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα ένα ταμείο για αυτή του είδους τη στρατηγική. Αυτό ξεπερνά τα όσα επιθυμούμε και τα όσα θέλουμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται ούτε να ζητήσουμε ένα επιπλέον προϋπολογισμό, ένα κονδύλι το οποίο να προχωρά πολύ πιο πέρα από τα όσα ζητά η έκθεση Γαρίγκα. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ενός τέτοιου κανονισμού. και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι από αυτό. Τώρα όσον αφορά ορισμένα στοιχεία συντονισμού, πρόκειται για τροπολογίες επί του κειμένου στο τρίτο τμήμα του κανονισμού όμως, ε, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα παράρτημα για τα θέματα περιβάλλοντος, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα καλύψουμε καλύτερα. Πάντως, πιστεύω πως γενικά συμφωνούμε για το ότι έχουμε 2.000 τροπολογίες. Δίνει την εντύπωση πως διαφωνούμε, πως δεν συμφωνούμε σε τίποτα, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Θα δούμε πώς θα το συζητήσουμε με τον συνεισηγητή ε, και πιστεύω ότι η θέση μας απέναντι στο Συμβούλιο θα είναι πολύ σταθερή. I'm just trying to wait till Martin Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν δεν έχει φτάσει ακόμη. Είμαστε σε κάπω δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε πότε θα έρθει ο Νίκολα Μάρτιν, σε πέντε λεπτά. Μάλιστα. Γιατί η Γραμματεία ήδη συνεργάζεται μαζί σας για τις συμβιβαστικές και Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε κάθε παραμικρό σχόλιο, γιατί εσείς οι συγητές θα μας δώσατε μια κάποια γραμμή για την πολιτική και για το μέλλον που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το τελευταίο χρόνο και πάνω από ένα χρόνο ως ομάδα εργασίας τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά μεταξύ μας. Και όλοι δραστηριοποιηθήκαμε και συμφωνούμε μαζί σας όσον αφορά την γενική κατεύθυνση της πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την κατεύθυνση αλλαγής ε, για τις πολιτικές. Δεν θα είναι εύκολο σε κάθε περίπτωση. Γιατί από ό,τι θυμάμαι στις συζητήσεις μας για το στατικικό πλαίσιο Νομίζω πως είχαμε σκεφτεί αρκετά νωρίς τα θέματα αυτά όσον αφορά το παράτημα ή τις κατεξουσιοδότης και όλα αυτά είναι σύμφωνα με το, τις συζητήσεις μας και την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Ίσως να είναι μια συμβιβαστική λοιπόν που μπορούμε να προτείνουμε. γιατί είναι σύμφωνα με αυτό που σκεφτόμασταν. Ξέραμε ότι θα χρειαζόμασταν κάτι πιο ευέλικτο και πιο εύκολο να αλλάξει, ώστε να βοηθήσουμε τα κάτι μελη και τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τον περίπλοκο χαρακτήρα των πολιτικών αυτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με όλε αυτές τις χιλιάδες τροπολογίες λοιπόν φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν συμβιβαστικέ που θα διατηρήσουν ωστόσο τη συνοχή τη πολιτική αυτή. και σε αυτό θα ήθελα να παραμείνουμε. Να όσοι θέλουν να φύγουν Α φύγουν. Εγώ θα μείνω να περιμένω τον Νικόλα Μάρτιν, αν θέλουν και οι συγκητές να μείνουν. Ε, κατά τα άλλα, κλείνουμε τη συμπροηνή μα συνεδρίαση, γιατί τα αποχηματινά θέματα δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει οι κατάλληλοι άνθρωποι εδώ. Ε, οι φαν του του Νίκολα Μάρτιν να μείνουν, οι υπόλοιποι φεύγουν, τέλος συνεδρίαση. και δεν θα χρειαστούμε και διερμηνήσει. Τέλος τη συνεδρίαση. Πρέπει να βαρέσω και το σφυράκι μου.